Ε, good Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συναδέλφοι. Θα δώσω ένα χρονικό περιθώριο στους συναδέλφους, στους φίλους, έτσι ώστε να φορέσουν τα ακουστικά τους. Να βρούνε ποια γλώσσα θέλουν να ακούσουν. Μπορείτε να δείτε δίπλα στον αριθμό της κάθε γλώσσας την γλώσσα να αναγράφετε με τον κωδικό της. Θα συνεχίσω να μιλάω έτσι ώστε να μπορέσετε να βρείτε κι εσείς ο καθένας στο κανάλι όσοι δεν το γνωρίζετε. Σας υπενθυμίσω ότι... Ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία για την ε, μνήμη των ε, βραβευθέντων αλλά και για να αναφέρουμε τα ονόματα των ε, παλαιότερων βραβευθέντων, το ε, Φόρουμ Σιμών Βέιλ, για να τιμήσουμε όλα τα ονόματα, όλες τις προσωπικότητες που έχουν βραβευθεί με το βραφείο Ζαχάροφ. Βλέπετε, γύρω μου σήμερα 12 βραβευθέντες με το βραβείο Ζαχάροφ. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι όλοι γνωρίζουμε πως είναι πολύ περισσότερος, πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός εκείνων που έχουν ε, που, οφείλουν που οφείλουμε να τιμήσουμε με το βραβείο Ζαχάροφ, που αξίζουν το βραβείο Ζαχάροφ, όλοι αυτοί οι πολίτες, οι εκατοντάδες εκατομμυρίων πολίτες σε όλο τον κόσμο που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τον αγώνα και για το παράδειγμα που δίνετε και σε εμά, σε όλους εμάς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, εδώ βρίσκομαι μπροστά σε όλους εσάς που έχετε υποφέρει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά που εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε δεδομένα. Και συνειδητοποιώ ότι πρέπει να δείξουμε πολύ μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνη τα επόμενα χρόνια, στο μέλλον, πολύ περισσότερη στράτευση και ενεργητική συμμετοχή στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο. Εσεί είσαστε εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών, αγωνιστέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφοι και δικηγόροι άνθρωποι που έχετε σηκώσει, υψώσει τη φωνή εκ μέρους όλων εκείνων που δεν έχουν φωνή. Και υποφέρατε γι' αυτό. Ταλαιπωρηθήκατε πολύ για τα ιδεώδη σας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι το προφανές για μας, αλλά όχι για, την κάθε, για το κάθε διδακτορικό καθεστώς, ότι δηλαδή έχει το δικαίωμα στην ζωή και την σωματική ακαιρεότητα ο κάθε άνθρωπος. Ταυτόχρονα όμως έχει και δικαίωμα στην ελευθεροτυπία, την ελευθερία του, ε, της συνειδήσεως, της σκεφτικής συνειδήσεως, της σκέψης, της εκφράσεως. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε παρά να έχουμε δικαιώματα από τους λίγους και μόνο για τους λίγους. Δεν μπορούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρούμε ως δεδομένη τη, δεδομένες ελευθερίες και να επαναπαυόμαστε. Όσοι έχουν αναμνήσεις ακόμα τις, τους πρόσφατου παρελθόντων μας ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει ελευθερία. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να είναι κανείς ε, καταπιεσμένος, να αντιμετωπίζει κατασταλτικά καθεστώτα, να βρίσκεται στο σκοτάδι και ταυτόχρονα να ζητεί το φως και να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον. Οι βασικές αξίες στις οποίες εμείς προάγουμε δεν είναι ευρωπαϊκές αξίες, είναι οικουμενικές αξίες του ανθρώπου. Και ισχύουν για τον κάθε ένα, για την κάθε μία σε ολόκληρο τον κόσμο. Επαναλαμβάνω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι όλοι μας αγωνιζόμαστε για οικουμενικές αξίες. Αγαπητοί φίλοι, ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συνάντηση σήμερα. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη έναντι των ε, βραβευτέντων με το βραβείο Ζαχάροφ. Δεν ε, ε, θέλουμε να πηγαίνουμε μόνο από τη μία εκδήλωση απονομής στην άλλη δεν θέλουμε να περιοριστούμε μόνο σε αυτό και αυτό είναι προσωπική μου πεποίθηση και γι' αυτό αποφασίσαμε να θεσπίσουμε το δίκτυο, την πλατφόρμα εκείνη δηλαδή, που θα επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, την ε, ε, γνώση, την απόκτηση της, ε, την αγαλλαγή εμπειριών, ο ένας από τον άλλον μπορούμε να μαθαίνουμε, μπορούμε εμείς να μαθαίνουμε από εσά και έτσι να οικοδομήσουμε πάνω στη δική σας τη στράτευση, πάνω στη δική σας την εμπειρία ανεκτήμητης αξίας εμπειρία για ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό βέβαια με δεδομένο ότι αλλάζει ταχύτατα ο κόσμος στην Ανατολική αλλά και στην Νότια γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζούμε την ιστορία που αλλάζει και εδώ βεβαίως περισσότερο από ό,τι ποτέ πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της οικοδόμησης των νέων καθεστώτων η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μόνο ένα συνονθήλευμα, ένα συνάθροισμα των εθνικών συμφερόντων, των συμφερόντων δηλαδή των κρατών μελών. Είναι πολύ περισσότερο από αυτή την απλή πολιτική. Είναι κοινέ πεπιθήσει. Είναι κοινέ υποχρεώσει. Δεν μπορώ να εκφράσω πιο εύγλωτα από ότι αν σου τσί όταν προσπαθούσε να πείσει τις κοινωνίες λέγοντας χρησιμοποιήστε παρακαλούμε τις δικές σας ελευθερίες για να προαγάγεται τις δικές μας. Έτσι έλεγε. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει σενάριο πολιτικής ε, με... μεταξέλιξης, μετάβασης. Κάθε χώρα πρέπει να βρει τη δική της λύση όπως συνέβη και με την ε, Πορτογαλία, την Ισπανία, την κεντρική ανατολική, ε, τις κόρες κεντρικής ανατολικής Ευρώπης, τη Σερβία τώρα τον αραβικό κόσμο. Δεν έχουμε ε, καμία θέση εμείς να δίνουμε διδάγματα και μαθήματα δημοκρατίας, αλλά μόνο να υποστηρίζουμε και να λαμβάνουμε έμπνευση από εκείνους που αποτελούν τον πραγματικό μοχλό της αλλαγής. Και είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, σκέψεων έτσι ώστε κάθε πολιτική μετάβαση να μπορεί να αντικατοπτρίζει τη βούληση των λαών. Και γι' αυτό το σκοπό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει έναν πληρέστατο διάλογο, έναν ε, ολιστικό διάλογο με την κοινωνία. Τα πολιτικά κόμματα η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να έχει εγγυημένο δικαίωμα να εκφράζεται, να εκφράζει τα αιτήματα και τις απαιτήσει για την ε, αλλαγή και για το ρυθμό της αλλαγής. Δεν θα πρέπει σε αυτό να αντιμετωπίζει τον εκφοβισμό, την τρομοκρατία των αρχών, όπως συμβαίνει σε πολλές ακόμη δυστυχώς περιοχές του κόσμου. Όπως πρέπει να υπενθυμίσω. Φερρυπίν Φιβέτ. με τη βία η καταστολή κατά των διαδηλωτών, με αδικαιολόγητες νομικές πιέσεις βάρος της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων, των θρησκευτικών ενώσεων ή όπως συμβαίνει στην ε, Συρία, τις ε, βίες καταστολές ή και στην Αίγυπτο ακόμη, οι ειδήσει που λαμβάνουμε είναι πάρα πολύ ανησυχητικέ. Αλλά από άλλες περιοχές του κόσμου είναι αρκετά ενθαρρυντικά τα νέα και ελπίζω ότι φερειπίνει αρχές στη Μιανμάρ πρώην Βυρμανία θα ε, τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για να προχωρήσουν στις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για πραγματικό δημοκρατικό καθεστώς, ανώθευτες και δίκαιες εκλογές και εγγύηση βασικών ελευθεριών. Όπως ξέρετε, η Αούγκ Σαν Σουτσί, με το βραβείο Ζαχάροφ, τις οποίες τα λόγια σας ανέφερα και νωρίτερα, και η Εθνική Ένωση και τη Δημοκρατία, της οποίας ηγείται, βρίσκονται στην πρωτοπορία αυτού του αγώνα. Η πιο σημαντική βέβαια για μας ερώτηση είναι πώς μπορούμε να συμβάλλουμε για τη μετάβαση προς τη δημοκρατία. Πρώτα, από όλα με τις κοινέ μας αξίες, με το συμφέρον του πολίτη ως επίκεντρο των δράσεών μας. Και γι' αυτό το Κοινοβούλιο επιμένει για περισσότερους πόρους στην στήριξη της, παρακο... της επιτήρησης εκλογών ή της επιτήρησης διαδικασία για την οικοδόμηση των δημοκρατικών θεσμών της κοινωνίας των πολιτών, των, των πολιτικών κομμάτων σε χώρες που βρίσκονται στη μετάβαση αυτή. Δεύτερον, μέσω πρόθεσμα, η, ε, η οικοδόμηση οικονομικής ευημερίας είναι ο μόνος όρος για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας, για τη βιωσιμότητα της δημοκρατίας, γιατί συνήθως είναι ένα απλό και φυσιολογικό πρόβλημα μία-δύο ε, χρονιές, ένα-δύο έτη μετά την ε, επανάσταση, τη μετάβαση προς τη δημοκρατία, να τίθεται ένα αμφιβόλο το μέλλον και η ευημερία μιας χώρας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιληφθούμε και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις νεότερες γενναίες, γιατί πρέπει να τους δώσουμε σαφείς προοπτικές για το μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να υποστηρίζει το ε, μέλημα ή ενίσχυση ή τα κονδύλια να αποβλέπουν σε αυτόν τον στόχο. Τρίτον και μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την οικοδόμηση ενός ενιαίου μοντέλου, ενός μοντέλου αντίστοιχου με αυτό που είχαμε στις χώρες μας. Πιστεύουμε σε αυτό το μοντέλο και εκ προσωπικής εμπειρίας μπορώ να σας πω ότι για διαφόρους λόγους και είτε πρόκειται για τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, αλλά παλαιότερα τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη, είμαι πεπισμένος ότι η σταδιακή ολοκλήρωση των γειτόνων μας μεταξύ τους, αλλά και η ενσωμάτωσή τους ή η ολοκλήρωση με τα δικά μας κράτη μπορούν να αποτελέσουν έναν πολύ ασφαλή δρόμο για τη δημοκρατία. Φυσικά δεν μπορούμε να προσφέρουμε ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε χώρα που βρίσκεται στη γειτονία μας. Πλην όμως μπορούμε να αποτελέσουμε εμείς ένα φάρο ειρήνης και ευημερία με την οικοδόμηση ενός τέτοιου χώρου και πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια αμοιβαία υποφελής σχέση. Είμαστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και κυρίε και κύριοι, επιτρέψτε μου ολοκληρώνοντας να πω δύο λόγια για τη σημασία της τεχνολογίας και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ως ε, τρόπο υποστηρίξη τη κοινωνία των πολιτών. Στη δεκαετία του 80. Η αλληλεγγύη η στάση της έναντι της, ε, και η έκφραση θέσεων σε σχέση με την, ε, με, με, τις, με την κατάσταση της δημοκρατίας και μέχρι και την άνοιξη του 1989 για μας, τι μέσα είχε, είχε τον πολύγραφο, είχε την ε, ε, μηχανή και είχε τον λόγο. Αυτή ήταν η Σολιδαρνόσκ της Πολωνίας. Τώρα όμως αυτοί οι νέοι, αυτά τα κινήματα έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ίντερνετ. Πολύ καλύτερα, αρκετά καλύτερα, αλλά και πιο επικίνδυνα μέσα. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους ε, ε, από τους γραφειοκράτες με το γραφείο Ζαχάροφ αξιοποιούν εν μέρη τις δυνατότητες αυτών των μέσων. Ο Τούτζα στην ε, Κίνα, επί παραδείγματι, είναι ένας από αυτούς τους ε, ακτιβιστές που δυστυχώς δεν είναι σήμερα μεταξύ μας, αλλά αξιοποιεί με τα μπλοκ του ε, και την παρουσία του μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, τη σύγχρονη τεχνολογία. Το ίδιο συμβαίνει και στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης. Υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να, την αξιοποιήσουν τεχνολογία για την αναζήτηση της ελευθερίας. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν για την ε, λογοκρισία, για τον έλεγχο, για την καταστολή. Γι' αυτό δεν είμαστε πάντοτε βέβαιοι ότι η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στις χώρες μας, στις χώρες σας σήμερα είναι καλύτερη φέτος από ότι το 80 στη δική μου τη χώρα, στη δεκαετία του 80, που δεν είχαμε τα τεχνολογικά αυτά για να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Δεν είμαι σίγουρο ότι τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Πρόκειται όμω για μια νέα πρόκληση. Πρόκειται για μια πρόκληση ε, για όσου αγωνίζονται για την προαγωγή και την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι οι μεγάλε εταιρείε έχουν και ιδιαίτερε ευθύνε, οι μεγάλε πολυεθνικέ. Επί παραδείγματι, έχουν ευθύνη. Έχουν την ευθύνη να συμβάλλουν σημαντικά στην ε, ε, εξασφάλιση του δικαιώματος, στην έκφραση και την ελεύθερη σκέψη. Ταυτόχρονα έχουν την ευθύνη να μην καταστούν υποχείρια των καθεστώτων καταστολής. Αγαπητοί φίλοι, την Αραβική Άνοιξη μερικοί την χαρακτήρισαν ε, επαναστάσεις του ίντερνετ. Αλλά δεν ήταν ούτε το facebook ούτε το twitter εκείνο το οποίο έριξε, ανέτρεψε τα ε, κατασταλτικά καθεστώτα. Όχι, το πνεύμα της ελευθερίας, το πνεύμα του ανθρώπου που αναζητεί ένα καλύτερο, μια καλύτερη ζωή ήταν αυτό που τα κατάφερε. Και αυτό είναι ακριβώς το πνεύμα το οποίο ε, κερδίζει αυτόν τον αγώνα. Τα λόγια, ο λόγος παραμένει πολύ ισχυρό όπλο. Η Μπεναζίρ Μπούτο, και πρέπει να σας παραθέσω τα λόγια της, είχε πει το εξή κάποτε. Έναν άνθρωπο μπορεί να το φυλακίσει κανείς, αλλά όχι μια ιδέα. Έναν άνθρωπο μπορεί να τον εξορίσει κανεί, αλλά δεν μπορεί να εξορίσει μια ιδέα. Έναν άνθρωπο μπορεί και να τον σκοτώσει κανείς, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει μια ιδέα. Και η ιδέα, η κοινή σε όλου μας, είναι η ιδέα, το ιδεώδες τη ελευθερία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Uh, Αν μου επιτρέπετε, θα δώσω το λόγο τον κύριο Σέργε Κοβάριεφ. Δύο χρόνια πριν συζητούσαμε με τους βραβευθέντες του βραβείου Ζαχάροφ και μιλήσαμε για ένα μνημείο, για τη δημιουργία ενός μνημείου, για, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ε, δίκτυο των βραβευθέντων με το βραβείο Ζαχάροφ. Και με την πρώτη προεδρία στην ιστορία μας θα ήταν κάτι τέτοιο, μία μνημειώδης χειρονομία. Γι' αυτό, αυτό συζητήσαμε με τον κύριο Κοβάριεφ. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω αγαπητέ φίλε από τη Ρωσία να μας μιλήσετε. Εσείς είσαστε ο συνειδητής μίας ρωσικής μη κυβερνητικής και από το 1988 προβάλλει την αλήθεια ως προς την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Αυτό είναι ύψης της σημασίας για μας. Παράλληλα, αγαπητέ φίλε Κοβάρεφ, δημιουργήσατε την πρώτη ένωση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σοβιετική Ένωση το 1969, αν δεν κάνω λάθος. 68 το 68. Ε, μπορούμε να προωθήσουμε και ένα διάλογο επί του θέματος. Λοιπόν, βραβείο Ζαχάροφ 2009. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι και η Λουτμίλα Αλεξέγεβα βραβεύθηκε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λυπάμαι ο κύριος Όλοφ δεν μπόρεσε να έρθει εδώ, αλλά θα ήθελα να καλωσορίσω τουλάχιστον εσάς τους δύο. Ξέρουμε ότι δίνεται αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω από 40 χρόνια. Κύριε Κοβάλευ και Αλεξέγεβα, έχετε το λόγο. Ο κύριος Κοβάλευ και μετά σε εσάς. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για το σαφή και εντυπωσιακό σας λόγο και την εισήγησή σας. Σε σχέση με τον φίλο ολεκολόφ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ για ε, τεχνικούς ας το πούμε λόγους και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μίνσκ, στο δικαστήριο του Μίνσκ και νομίζω ότι θα γίνει λόγος για την δίκη αυτή σήμερα. Αρχίζω λοιπόν με την παρέμβαση, την ομιλία μου. Η διάσκεψη αυτή φέρει το όνομα Ζαχάροφ. Είναι απόλυτα λογικό κάτι τέτοιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε την απόφαση της δημιουργίας του βραφείου Ζαχάροφ, γι' αυτό και η διάσκεψη φέρει αυτό το όνομα. Και μπορούμε να πούμε ότι το πνεύμα του ε, Ζαχάροφ μας ε, διαπνέει και εμάς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα από αυτό να σας πω μερικά λόγια. Ο Ζαχάροφ είχε προωθήσει μια καθαρά ρεαλιστική πολιτική και πάντα θέλησε να κινηθεί πέρα από αυτή τη ρεάλ πολιτικ. Αυτή ήταν η βασική του ιδέα και επιθυμία. Διότι η ρεάλ πολιτικ δεν απέδωσε κατέδειξε τα όρια της και ήταν επικίνδυνη για όλους μας. Η μεγάλη πλειοψηφία ή μάλλον όλοι οι βραβευθέντες του βραβείου Ζαχάροφ εκπροσωπούν χώρες όπου τα πράγματα ε, δεν βαίνουν καλώς. Σπάνια εκπροσωπείται κάποιος από το δυτικό κόσμο. Όμως οι καθολικές αξίες αφορούν όλους τους πολιτικούς που σέβονται ή δεν σέβονται τον εαυτό τους. Μιλάμε για καθολικές αξίες που είναι απότοκες της ευρωπαϊκής πολιτισμικής βάσης. Πρόκειται για καθολικές αξίες αλλά απορρέουν και από την εξέλιξη του ευρωπαϊκού ευρωπαϊκού πολιτισμού και θα μπορούσα να προσθέσω του χριστιανικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Άρα οφείλουμε να αναρωτηθούμε γιατί οι χώρες οι οποίες ε, καταξίωσαν αυτές τις αρχές δεν βρίσκονται εδώ ως βραβευθέντες. Γιατί δεν βρίσκονται όλοι, γιατί δεν είναι όλοι παρόντες. Γνωρίζετε πώς έχει η κατάσταση παγκοσμίω υπάρχουν πολλά αιμοσταγή καθεστώτα και δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα ότι η κρίση που πλήττει τον αλληλένδετο κόσμο μας δεν είναι οικονομικού χαρακτήρα. Είναι μια παγκόσμια κρίση ηθικών αξιών, ιστορικής και πολιτικής υφής. Πρόκειται για ένα είδος κοινωνικού δαρβινισμού και πολλές φορές με την πολιτική του ο Νικολό Μακιαβέλη άνοιξε το δρόμο σε μακιαβελική, οι μακιαβελικές τακτικές. Και γι' αυτό θεσπίστηκε και το βραβείο Ζαχάροφ. Κύριο μας μέλημα ήταν να προασπίσουμε τις ανθρώπινες αξίες ανά τον κόσμο. Ο, κόμος, ο κόσμος όμως ξέχασε αυτή την πάγια θέληση του Ζαχάροφ. Θα ήθελα να σας ε, δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα με τον μεγάλο μου φίλο. Είμαστε υπέρμαχοι της Realpolitik και κάποια μέρα συζητούσαμε μεταξύ μας για τη διάσκεψη της Γιάλτας. Οι χώρες που νίκησαν και η Γερμανία που ιτήθηκε. Μιλούσαμε για τις ε, χώρες της Συμμαχίας και επήλθε μία συμφωνία. Μιλούσαμε για 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους που έδωσαν τη ζωή τους. Αυτό ήταν κάτι το τερατώδες απότοκο του οποίου ήταν και η διάσκεψη της Γιάλτας και ο φίλος μου μου είπε «Έχεις δίκιο». Αλλά αν ήσουν εσύ στη Γιάλτα, τι θα είχες κάνει εκείνη την εποχή. Τι απόφαση θα είχες λάβει. Με έφερε σε δύσκολη θέση αυτό το ερώτημα και κατάλαβα τι ήθελε να πει. Θα έκανα το ίδιο με αυτό που έκαναν οι Ρούσβελτ και Τσόρτσιλ έναντι του Στάλιν. Αυτό είναι το πιο τομερό στοιχείο της πραγματικότητας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά σε έναν κόσμο όπου μπορούμε να οργανώνουμε διασκέψεις τύπου Γιάλτα και όπου οι Ευρωπαίοι απέκτησαν την ελευθερία τους με αντίτιμο τη ζωή άλλων ανθρώπων. Ευρωπαίων. Και αυτό αντικατοπτρίζει και το βραβείο Ζαχάροφ. Νομίζω ότι είναι ο μόνο άνθρωπος που γνώρισα που εξέφραζε την αγανάκτησή του ανοιχτά ως προς τη δυστυχία των άλλων, των άδικων δικών και ζούσε, φαινόταν σαν να ζούσε το δράμα των άλλων. Αυτό καταδεικνύει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ήσυχα σε μια γωνιά του κόσμου χωρίς να κατανοούμε τον αλληλένδετο χαρακτήρα των ε, παγκοσμίων δρομένων. Δεν ήταν ο μόνος που σκεφτόταν έτσι. Ο Νίλς Μπορ και πολλοί άλλοι σκέφτονταν κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορώ να προβώ σε έναν απογραφικό κατάλογο αυτών που σκέφτονταν έτσι ο Νίλς Μπορ, ο Άλμπερτ Άινστάιν και πολλοί άλλοι. Έχω κατά νου και πολλούς άλλους Προσπαθώ να σκεφτώ και ένα το όνομα ενός Άγγλου φιλόσοφου που γνωρίζω πολύ καλά και θα, θα θυμηθώ το όνομά του. Θα όφιλα να αναφέρω και τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ που ήταν υπέρμαχη αυτού του νέου τρόπου σκέπτεσθε ναι, Bertrand Ράσελ, το θυμήθηκα, το θυμήθηκα. Λέει ο βραβευτής ο κύριος Κοβάλεφ. Ε, πρόκειται για τον Bertrand Ράσελ. Το όνομά του μου διέφυγε προς στιγμή. Όλοι έλεγαν το ίδιο επί της ουσίας. Δηλαδή μιλούσαν για ένα καλύτερο μέλλον, όπου οι μεγάλες καθολικές αξίες θα ισχύουν εν της πράγμαση και θα αποτελέσουν την πραγματική βάση της πολιτικής, της πολιτικής μας. Ο καθένας βεβαίως είχε τη δική του ερμηνεία των πανανθρώπιων πανανθρώπινων αξιών και νομίζω ότι ο Αντρέι Ζαχάροφ σκέφτηκε εις βάθος αυτό το ζήτημα. Δεν είναι ούτε ο τόπος ούτε ο χρόνος να το συζητήσουμε αυτό το θέμα εις βάθος. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σκέπτηση, τον τρόπο σκέπτεσθε του Ζαχάροφ και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε πολύ καλά προς αυτή την κατεύθυνση. Η ολοκλήρωση της Ευρώπης ήταν ένα δύσκολο μονοπάτι γεμάτο αντιφάσεις και προσκόμματα και το πέρασμα από την Οικονομική Ένωση σε μια πολιτική ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν έμφυτη από αντιφάσεις. Θυμάμαι και το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Όλες αυτές οι χέριες είναι αναπόφευκτες. Όμως υπάρχει δρόμος υπέρβασης όλων αυτών των δυσχεριών. Τη στιγμή που ζούμε σε έναν κόσμο όπου μια, χειροσύμα και ένα ανακασάκι ε, είναι αναπόφευκτα και όπου υπάρχουν διασκέψεις τύπου Γιάλτας, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιόν μας. Νομίζω ότι αυτή η εξαίρετη πρωτοβουλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή η δημιουργία ενός δικτύου για τους βραβευθέντες είναι ένα μικρό βήμα γεμάτο ελπίδες και που κινείται προς την καλή κατεύθυνση. Νομίζω ότι αυτή η κοινότητα των βραβευθέντων, Ζαχάροφ, θα πρέπει να συνέρχεται μία ή δύο φορές το χρόνο για να συζητά Ίσως θα έπρεπε να προβλέψουμε και μία μόνιμη υποδομή γιατί μας διέπουν αυτά τα ιδεώδη τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ευχαριστούμε κύριε Κοβάλευ. I would like to ask for taking floor, Madame Ludmila Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λουμπμίλα Αλεξέγεβα. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ευτυχής και υπερήφανη που βρίσκομαι εδώ. Που βρίσκομαι εδώ με τους άλλους βραβευτέντες, με το βραβείο Ζακχάροφ, βραβευτέντες από διαφορετικές χρονιές και πολλές χώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε Μπουζέκ για αυτή τη μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να διαβάσουμε ο ένας για τον άλλον, αλλά για να μπορέσουμε να συναντηθούμε και να συζητήσουμε μεταξύ μας. Να μιλήσουμε δηλαδή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και για το έργο μας. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ευτυχής που είμαστε όλοι ενωμένοι με την ιδέες και το όνομα του Αντρέη Ζακάρο και ας προερχόμαστε από πολλές άλλες χώρες, διαφορετικές χώρες. Είναι συγχρονός μου, αν μπορώ να το πω έτσι, ένας μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος άντρας, μεγάλη προσωπικότητα που τέτοιες δεν φτιάχνει κάθε γενιά. Για όλους τους βραβευτέντες με το βραβείο Ζαχάροφ, αλλά όχι μόνο για αυτούς αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που συνεργάζονται, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στις χώρες μας. Ο Αντρέι Ζαχάροφ είναι ένα ιδανικό, κάτι που είναι αδύνατον να γίνει χειροπιαστό, να το φτάσουμε τουλάχιστον, αλλά είναι κοινό ιδανικό. Πέρυσι βραβεύτηκαν ο συνάδελφος Σεργέη Κοβαλιέφ, εγώ και ο Αλιέγ Ορλόφ, που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εδώ. Είναι ο επικεφαλής της οργάνωσης Memorial, προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι στο Μίνσκ σήμερα, διότι εκεί διεξάγεται η δίκη σήμερα Ενό συναδέλφου του Αντρέη Μπιλιεύσκη που είναι επικεφαλής της ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λευκορωσία. Αυτή η οργάνωση λοιπόν προσπαθεί να βοηθήσει όλους εκείνους που αγωνίζονται να εξασφαλίσουν η Λευκορωσία να γίνει δημοκρατική χώρα με κράτος δικαίου να γλιτώσει από το ζυγό της δικτατορίας με ειρηνικά μέσα. Ο Πελιεύσκη λοιπόν καταδικάστηκε σήμερα για πέντε έτη φυλάκισης. Ελπίζω λοιπόν, ότι θα καταβάλουμε όλοι οι προσπάθειες ώστε από κοινού μάλιστα, ώστε οποιαδήποτε και αν ήταν η απόφαση του δικαστηρίου ο Παλιεύσκη να μπορέσει να απελευθερωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τους βραβευτέντες, επισκέπτες μας και προσκεκλημένους ε, να λάβουν το λόγο σιγά σιγά. Η κυρία Γκαζάρη. Αλγερινή δημοσιογράφος από τη Βόρεια Αφρική. Πολύ συμβολική προέλευση για όλους μας. Στο, στο βιογραφικό σας λέει ότι αγωνιστήκατε για τα γυναικεία δικαιώματα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά για μένα αυτά είναι τα ίδια πρέπει να σας πω. Βεβαίως, οι γυναίκες είναι άνθρωποι και τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεπώς ανήκουν σε όλους. Ε, βραβευθήκατε το 1997. Ήσασταν μωρό τότε, <laughs> λέει ο πρόεδρος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους όσους βρίσκεστε εδώ σήμερα. Μιλάμε πάρα πολύ για τους βαβραφέντες με το βραβείο Ζαχάροφ. Είναι καλό πράγμα βέβαια αυτό. Αλλά νομίζω ότι η διομορφία της σημερινή στιγμής είναι ότι μιλάμε για την ώρα Ζαχάροφ. Μιλάμε για την παγκοσμιότητα των δικαιωμάτων για την παγκοσμιότητα των αξιών, των αξιών της δημοκρατίας. Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσα πράγματα δηλαδή τα οποία μας ενώνουν στον αγώνα μας, στις συναντήσεις μας, στις προσπάθειές μας. Χρον, πρέπει να μιλήσουμε όμως και για την παγκοσμιότητα των πρωταγωνιστών και των δράσεων. Όταν μου δόθηκε το βραβείο Ζαχάροφ το 97, δεν ήταν επειδή είχα κάποια προσωπική ιδιομορφία. Ε, είχε σχέση με την κατάσταση στη χώρα μου, με τον αγώνα της, ε, για την ανεξαρτησία από τη σκλαβιά ε, που υφίστανται οι άνθρωποι μετά την απεικιοκρατία. Πολλά πράγματα ήταν ανυπόφορο και πολλοί φίλοι της Αλγερίας ε, στράφηκαν προς την Αλγερία για να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των πρωταγωνιστών της κοινωνίας των παλιτών της Ευρώπης. Μιλάω για, βασικά για ΜΚΟ που αγωνίστηκαν στο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα προσπάθειες γίνανε από οργανώσεις ευρωπαϊκές, πολιτικές, θρησκευτικέ, ε, να βοηθήσουν τους Αλγερινούς για να υλοποιήσουν μια πρόταση που ήταν φάρος κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας, δηλαδή την κυριαρχία του πολιτικού κατά του στρατιωτικού. Ήταν ένας αγώνας που δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε για πολύ χρόνο η κοινότητα σαν Legion μας βοήθησε να ενωθούμε. Δηλαδή από όλα τα κόμματα, σοσιαλιστές, δημοκράτες, μουσουλμάνοι, όλοι ενωθήκαμε γύρω από μια πρόταση πολιτικής σύμβασης. Όλα αυτά δεν είναι ξέμακρα, διότι το δημοκρατικό ζήτημα είναι η στιγμή υπέρτατη, είναι η στιγμή του αγώνα των αφρικανικών, βορειοαφρικανικών χωρών. Είναι ο αγώνας αυτών που έχουν βραβευτεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό επιδιώκουμε, ένα πολιτικό συμβόλαιο, ένα κοινωνικό συμβόλαιο να υλοποιηθεί στις χώρες μας αλλά και παγκόσμια. Και σύμφωνα απόλυτα με αυτό το οποίο ελέγχθη πριν από μένα, δηλαδή ότι η δημοκρατία και η παγκοσμιότητα είναι ένα σύνολο και ακριβώς πάνω σε αυτό το σύνολο, σαν συναλλαγές γύρω από αυτό το σύνολο βρίσκουμε το μήνυμα του διαλόγου μας και της συνάντησής μας. Δηλαδή αμοιβαία λέει ο ένας τον άλλον πράγματα τα οποία καμιά φορά είναι δυσάρεστα. Όταν μου δόθηκε το βραβείο το 1997 ένας αντίπολός μου πολιτικός στην Αλγερία μου είπε η ελευθερία του πνεύματος είναι πόσες διαιρέσεις. Όχι, δεν έχουμε πολλές διαιρέσεις. Γιατί, γιατί πιστεύουμε βέβαια στις διαιρέσεις, είναι θετικό πράγμα, αλλά αυτό στην πολιτική υλοποίηση. Συμβολικά όμως ε, δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μιλάω μόνο εγώ αλλά επανερχόμαστε στη σημερινή στιγμή μιλώντας για την Αραβική Άνοιξη. Είναι αγώνες που γίνανε μέσα στη μοναξιά. Έχουμε εδώ μάρτυρες αυτών των προσπαθειών δεκαετίες, χωρίς καμία υποστήριξη δεν αγωνιζόντουσαν. Και ε, υπήρχε και η εντύπωση ότι με τα ΜΜΕ ε, θα επιληθούν όλα υποστηρίζοντας κάτι χωρίς περιεχόμενο χωρίς υλοποίηση, παρά τα λάθη, όπως τα λάθη της κυρίας Μισελ Αλιομαρή όταν πρότεινε την αστυνομία της. Δεν ήταν ε, λεκτικό λάθος, ήταν ε, ε, μια διατύπωση η οποία αποκάλυψε τις ακριβείς σχέσεις μεταξύ των κρατών και των κρατών μας. Είμαι σκληρή στη διατύπωσή μου, αν θέλετε, στην τοποθέτησή μου για ορισμένους ανθρώπους. Ε, το γεγονός ότι μου δόθηκε το βραβείο Ζαχάρο πιθανότατα μου, σώθηκε, μου σώσανε τη ζωή. Αλλά αφού μου σώθηκε η ζωή, ε, μου δίνει τη δυνατότητα να διατυπώσω τις απόψεις μου. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα συγκεκριμένο όταν οι άλλοι ε, συνυπήκοοι μου, συμπολίτες μου δεν έχουν ε, τη δυνατότητα να διατυπώσουν την άποψή τους. Εγώ συνεπώς διατύπωνα μια πλειοψηφία μεν, αλλά μετά έρχεται μία αντιπροσωπεία της, από την Ευρώπη η οποία λέει ότι ξαφνικά υπάρχει μία πνοή δημοκρατία στην Αργερία. Μα δεν ήταν καθόλου ξαφνικά. Υπάρχει μία αντίφαση, ε, πράγμα το οποίο μας αναγκάζει καμιά φορά να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και να χάνουμε την πίστη μας. Αυτά ε, ε, είναι σημαντική δέσμευση του κάθε πολίτη στη δημοκρατία πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην υπόσχεση και στην κοινή ελπίδα. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία στο πνεύμα, πίστη στην πολιτική δράση και παγκοσμιότητα με την έννοια ότι και οι δικτάτορες δεν μπορεί ε, να βασίζονται στις διαιρέσεις για να επιβάλλουν τη στρατιωτική τους κυριαρχία αλλά και οικονομικά, ε, η οικονομική πτυχή είναι πραγματικά προσδιοριστική και θα τελειώσω για, και με συγχωρείτε για την αταξία της παρέμβασής μου, αλλά πρέπει να σας πω ότι φοβάμαι ότι αν ανάμεσα στη συμβολική χειρονομία αναγνώρισης ενός αγώνα οπουδήποτε στο πλανήτη και την αναγνώριση της οικονομικής και πολιτικής δράσης καθημερινά ε, η απόσταση ε, επιδεινωθεί φοβάμαι ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε Ισπανούς ε, που θα επιβραβεύονται Ιρλανδούς διότι και θα χρειαστεί να ξανααγωνιστούμε στην Ευρώπη για τις ελευθερίες, φοβάμαι στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία μου, λέει ο Πρόεδρος. Βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα λόγια σας, χωρίς να είμαστε πάντα απεσιόδεξοι βέβαια. Βέβαια θα λάβουμε υπόψη τα λόγια σας. Και τώρα έχουμε τον τιμηθέντα το 2006 με το βραβείο Ζαχάρεφ, Αλεξάνδρ Μιλίνκεβιτς. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι. Με χαρά είμαι εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση. Ξέρω ότι είναι πολύ σημαντική συνεδρίαση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του φόρουμ που μας επέτρεψαν όλοι μαζί να συναντηθούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας γιατί ενωμένοι είμαστε πολύ πιο ισχυροί. Όταν καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να ζούμε ελεύθεροι έστω και αν είμαστε σε διαφορετικές υπήρους, διαφορετικές χώρες. Όταν είμαστε ενωμένοι είναι πολύ πιο ε, περιορισμένες οι δυνατότητες των δικτατόρων, δεν μπορούν να μας αγνοήσουν, δεν μπορούν να αγνοήσουν τις διεκδικήσεις μας και τις θέσεις μας. Συχνά, σε συνεδριάσεις όπως η σημερινή, με ρωτάνε οι παρευρισκόμενοι πότε θα φτάσετε και εσείς στο ιδεώδες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ε, πότε θα τα καταφέρετε και εσείς όπως και οι άλλοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σας πω. Δεν μπορώ να δώσω χρονικό ορίζοντα δηλαδή, αλλά ξέρω ότι θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το καθήκον μας. Στον αγώνα για τη δημοκρατία ξέρω ότι πολλές φορές ε, αλλάζουν και οι μόδες. Το 2000 μιλούσαμε με χρώματα στις επαναστάσεις. Της Σερβίας, ε, της Ουκρανίας, της Γεωργίας. Δίναμε χρώματα. Και έτσι δινόταν και ζωή στους αγώνες των ανθρώπων που πια είχαν αγανακτήσει, δεν ήθελαν να ζουν στις ίδιες συνθήκες και διεκδικούσαν τις ελευθερίες τους. Όταν όμως έφυγαν με επιτυχία αυτές οι ελευθερίες, είδαμε ότι δεν μπορούμε να αρκιστούμε σε αυτά και πρέπει να ετοιμάσουμε τις ε, κοινωνίες μας ώστε αυτές οι επαναστάσεις να αποβούν και χρήσιμες, ώστε να μπορεί να ξέρει και ο δημοσιογράφος πώς θα διατυπώσει το λόγο του σε όρους ελευθερίας. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι δεν αρκούν οι χρωματιστές αυτές, οι άχρωμες αυτές ε, επαναστάσεις. Όταν το 2001 εγώ ήμουν υποψήφιος για προεδρία στη χώρα μου, ήξερα ότι δεν θα τελειώσει εκεί ο αγώνας. Λέγαμε ότι θα πάμε σε εκλογές, λέγαμε ότι θα διεκδικήσουμε με την επανάσταση να βγει ο κόσμος στους δρόμους, να ζητήσει δημοκρατικά δικαιώματα. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν θαραλέοι όσοι βγήκαν στους δρόμους, γιατί ξέραμε ότι και θα, μας, ε, και θα ανοίξουν πύρα ανάντιον μας και θα ανοίξουν πύρα εναντίον μας και θα μας κατηγορήσουν ως τρομοκράτες. Τώρα στην Βόρεια Αφρική βλέπουμε να αναπτύσσονται αντίστοιχε επαναστάσεις με πολύ θαραλέους ανθρώπους. Έχω μεν ε, καταγωγή από την ε, Ευρώπη, αλλά έχω σχέσεις ιδιαίτερες με την Βόρεια Αφρική, γιατί είχα ζήσει τέσσερα χρόνια στην Αλγερία. Ξέρω ότι πολλές φορές ε, η Ευρώπη εκφράζει αμφιβολίες ως προς τα ε, κινήματα αυτά, λέγοντας ότι μα, ο κόσμος μπορεί να θέλει να ζει κάτω από τέτοια καθεστώτα δεκτατορικά, μπορεί να προτιμούν την τάξη και την ασφάλεια. Ξέρουμε ότι μια ένα αυταρχικό καθεστώς μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, αλλά δεν ισχύει αυτό και το βλέπουμε με τις επαναστάσεις αυτές ότι ο κόσμος διεκδικεί την ελευθερία του και ξέρουμε επίσης ότι δεν αποτελεί εγγύη σταθερότητα σε ένα αυταρχικό καθεστώς, σε ένα δικτατορικό καθεστώς γιατί ό,τι και να γίνει εν τέλει θα καταλήξει σε επανάσταση η χώρα αυτή. Άρα και εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι η πορεία αυτή της επανάστασης δεν είναι μία στιγμή στην ιστορία που αρχίζει και τελειώνει. Χρειάζεται και τη συνέχεια της, χρειάζεται όχι μόνο να δώσουμε τέλος στους δικτάτορες και εδώ αναφέρομαι τώρα στη χώρα μου, πρέπει να αποφύγουμε να επανεμφανιστούν οι Λουκασέγκο. Και σε αυτό χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να, είμαστε, να έχουμε την εγγύηση ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι είναι δημοκρατία. Και αυτό που διεκδικούμε μεταξύ άλλων είναι ο εξευρωπαϊσμός της χώρας μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάρη σε αυτό, γιατί τακτικές μπορεί να υπάρχουν, αλλά στρατηγική χρειάζεται πάνω απ' όλα για να μπορέσουμε να βγούμε από την κατάσταση αυτή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στις χώρες του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ, είτε πρόκειται για την Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, προβλήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Λουβιάννα Αλεξέγεβα το είπε, αλλά και ο κύριος Κοβάλεφ μόλις τώρα, ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι. Έχουμε δύο υποψηφίους ε, πρωθυπουργού κρατούμεν φυλακισμένου αυτή τη στιγμή στη χώρα μου, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πολλέ δίκε ει βάρο αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μίνσκ που βρίσκονται εν εξελίξη. Εχθέ ο εισαγγελέα ζήτησε πλήρη δίμευση περιουσιακών στοιχείων και πενταετή φυλάκιση για δημοσιογράφο, ο οποίο υποτίθεται ότι δεν πλήρωσε το φόρο του στον στο δικτάτορα, στο δικτατορικό καθεστώς. Ε, από πού θα έπρεπε να πληρώσει φόρο, δεν πληρώθηκε από κανέναν. ε, φορέα, απλώς ε, είχε βοήθεια από ανθρώπους ε, που τον στήριζαν στη, στον αγώνα του αυτόν. Και τώρα φαίνεται ότι κινδυνεύει να φυλακιστεί για φοροδιαφυγή. Παρακαλώ λοιπόν όλοι εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο, όσοι μας παρακολουθείτε και από το διαδίκτυο, επιδείξτε την αλληλεγγύη σε αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρουμε ότι η δίκη θα συνεχιστεί ακόμη. Έχουμε όμως ξεκινήσει μια εκστρατεία των λόγω δημοσιογράφων να τον προβάλλουμε ως υποψήφιο για το Νόμπελ Ιρήνη το 2012 γιατί του αξίζει να τιμηθεί για τους αγώνες του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Λευκορωσία. Θέλουμε την ελευθερία μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρου. Και τώρα παρακαλώ την κυρία Μπλάνκα Ρέιες συνειδρήτρια των κυριών με Και όπως γνωρίζετε, είχαμε να κάνουμε, από, με, ε, είχαμε να κάνουμε με μητέρες, παιδιά, αδελφές, φυλακισμένων. Το 2005 κερδίσατε το βραβείο ε, Ζαχάροφ και έχετε το λόγο. Πρόεδρε. Φίλοι, βαραβευθέντες, φίλοι, με την βράβευση των ε, γυναικών στα Λευκά του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω το θάνατο της Λάουρα Πογιάν που απεβίωσε λίγες μέρες πριν και η οποία ήταν υπέρμαχος των αντιρρησιών συνείδησης. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε την ειρηνική μας πορεία ως γυναίκες της Κούβας και θα τιμούμε τον αγώνα μας με, υπό την Βέρτα Σολέρ, η οποία και εκπροσωπεί τις γυναίκες στα λεφτά στα λευκά. Από το 2003 όταν την Μαύρη Άνοιξη η κυβέρνηση φυλάκισε 75 ακτιβιστές οι οποίοι ήταν κυρίως δημοσιογράφοι, αρχίσαμε να υπερασπιζόμαστε τους δικούς μας ανθρώπους με εκδηλώσεις, πορείες και στην Κούβα και στο εξωτερικό. Γιατί ξέραμε τι κίνδυνους διέτρεχαν οι φυλακισμένοι μας υπό το κουβανικό καθεστώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες παρατηρητών ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχουν 80 φυλακισμένοι αντιρρησίες. Α, αυτοί μας οδήγησαν να κινηθούμε σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες, να μπορούν να βγαίνουν και να μπαίνουν στη χώρα τους και να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους. Οι γυναίκες στα Λεύκα αποτέλεσαν την κορονίδα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα, χωρίς χρήση ιδεολογημάτων και θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε την ελευθερία στην Κούβα. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι μας υποστήριξε μια οργάνωση δημοκρατικά εκλεγμένη. Σας ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σας. Θα ήθελα να κινηθώ στους ε, δημοσιογράφους χωρίς σύνορα. Τους βραβευθέντες το, του 2005 έχουμε έναν εκπρόσωπο, τον κύριο Ολιβιέ Μπαζίλ και ξέρουμε ότι εκπροσωπείται μία μη κυβερνητική οργάνωση Μιλάτε για την ελευθεροτυπία που είναι ύψης της σημασίας μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας γενικότερα και του αγώνα υπέρ της ελευθερίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά ξαναβρισκόμαστε ως βραβευθέντες είτε στο Στρασβούργο είτε στις Βρυξέλλες, βεβαίως πρέπει να εκφράσουμε την πικρία μας, γιατί πολλές φορές λείπουν αρκετοί βραβευθέντες, όχι για λόγους υποχρεώσεων. Ο μοφαρίνας Λεπάγε και ο Σανσούκη. Και δυστυχώς μας μένει αυτή η πικρή γεύση, διότι δεν εκπροσωπούνται τέσσερις άλλοι βραβευθέντες από τους δημοσιογράφους χωρίς ε, σύνορα. Μέσα στα πλαίσια αυτών των ημερίδων περισυλλογής ε, καλείται πάνελιστ οι οποίοι προβαίνουν σε πολύ εύστοχες αναλύσεις αλλά μετά δεν περνάμε στη δράση. 15 χρόνια είμαι δημοσιογράφος και στα ευρωπαϊκά όργανα και βλέπουμε ότι μία μακρά ημέρα αρχίζει μόλις. Θα πρέπει να μας απασχολεί η συνοχή και η δράση. Συνοχή γιατί μιλάμε για την αραβική άνοιξη, αλλά παράλληλα κάνουμε έναν απολογισμό των δραστηριοτήτων μας εδώ και 20 χρόνια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για μια πολιτική που προωθήσαμε ως Ευρωπαίοι πολίτες. Χαιρετίζουμε λοιπόν την Αραβική Άνοιξη και τα ηλεκτρονικά μέσα αλλά βλέπουμε ότι και εδώ στο Κοινοβούλιο υπάρχουν ε, κείμενα που αντίκυνται σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, όπως η άκτα. Κάτι το οποίο πάντα μας λένε στους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα ότι δεν γίνεται κατανοητό εξαιρετικό το διαδίκτυο, το facebook, αλλά παράλληλα υπάρχει μία νομοθετικού τύπου αιμορραγία μέσω συμφωνιών οι οποίες είναι ιδιαίτερα δόλιες και επιζήμιες για την πληροφόρηση των πολιτών. Πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και συνεπείς. Ψηφίζουμε προτάσεις ψηφισμάτων, αλλά παράλληλα δεν μπορείτε να καταδικάζετε χώρες όταν δεν, τις δεν αντιμετωπίζετε θέματα ελευθεροτυπίας και ελευθερίας του εκφράζεστε στις δικές σας χώρες, δηλαδή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προωθήσουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, αλλά υπάρχει μεγάλη παλινοδία και οπισθοδρόμηση ως προς την ελευθεροτυπία και την ελευθερία του εκφράζεστε. Και εάν δεν προχωρήσουμε σωστά γιατί άκουσα ε, για την λευκή βίβλο σας, κύριε Μπούζεκ. Σημερίζομαι αυτή την ανάλυση που προωθείτε και που βλέπω στον τύπο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα χάσμα στο ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για υπεράσπιση δικαιωμάτων ελευθερίας του εκφράζεστε ιδιαίτερα ως προς τον ε, θρησκευτικό προσανατολισμό και μετά να μιλάμε για ένα ανάθεμα 25.000 ευρώ. Κανένας δεν είδε την έλευση της Αραβικής Άνοιξης. Ίσως αύριο θα πρέπει να δώσουμε το βραβείο Ζαχάροφ σε κατοίκους της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας. Βλέπουμε ότι δυστυχώς η ελπίδα χάνεται και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Μίλησα για συνοχή αλλά και για δράση. Εγκαινιάσαμε τον περίπατο Ζαχάροφ κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ωραίο. Χαιρόμαστε να, βλέπουμε το, να ακούμε το όνομα Ζαχάροφ στις Βρυξέλλες, αλλά αυτός ο περίπατος θα πρέπει να μας οδηγήσει στον οίκο Ζαχάροφ. Θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας έτσι ώστε σε αυτό το δίκτυο να συνεπάρξουν αυτοί που πιστεύουν και αυτοί που δεν πιστεύουν και τόσο πολύ. Πρόκειται για ένα δίκτυο συμβούλων, δημοσιογράφων, δικηγόρων και εδώ λαμβάνω υπόψη ε, εφημερίδες της Λευκορωσίας, της φίλης μας που μίλησε από πλευράς Αλγερίας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι βραβευθέντες δεν είναι μόνοι και όπως είπε η Σαλιμά, πολλοί δεν έχουν φωνή και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν στις Βρυξέλλες. Να μιλήσουμε ανοιχτά για shelter cities. Θα πρέπει να δούμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα shelter cities χρειάζονται, διότι πολλοί έπρεπε να ζήσουν ως νομάδες πολλά χρόνια, χωρίς να μπορούν να σταματήσουν. Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτού του είδους της πόλης και μέσω ηλεκτρονικών δικτύων τις προωθήσουμε, τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία υπογραμμίσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Θα αγωνιστούμε βεβαίως όλοι για αυτήν την μορφή που έχουμε πιστεύω για όλους σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι δεν ασφαλίσει κανείς και πουθενά και πιστεύω ότι εδώ συμφωνούμε τουλάχιστον όλοι στο Προεδρείο, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας επόψεις. Εάν θέλετε για μια πιο σύντομη παρέμβαση. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα αρκεστώ σε δύο σημεία γιατί αυτό που με, μας ενδιαφέρει είναι να λάβουμε υπόψη όλες τις διαστάσεις της ε, βράβευσης. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα προώθησαν ιδέες έμπρακτα που θα έπρεπε να προωθήσουμε ή τουλάχιστον να συζητήσουμε. Και κάτι άλλο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μας ζητούν δράση στον τομέα των θεμελιωδών ελευθεριών και πολλές φορές τα κράτη-μέλη δεν το προωθούν αυτό. Με βάση, μάλλον επικαλούμενη την αρχή της επικουρικότητας. Όμως η επικουρικότητα δεν μπορεί να αποτελέσει πρόσκομα, πρόσκομα κατά της έκφρασης της ελευθερίας και αυτό αφορά και τα ψηφίσματά μας σε σχέση με την Ουγγαρία και την ελευθερία στα ΜΜΕ της Ουγγαρίας. Επειδή ακριβώς ε, ακολουθήσαμε στεναρή στάση μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε γιατί οι Ούγγροι βρίσκονταν μέσα σε μία μαύρη τρύπα και δεν μπορούσαν να ε, υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Αυτό κάνουμε μετά το 89 για τις χώρες αυτές. Επίσης, επιγραμματικά και αποτινόμενος τους φίλους μας από τη ε, ε, Ρωσία θα ήθελα να πω ότι στον πορτογαλικό ε, τύπο μετά το θάνατο της Ελένα Μπόνερ, της Ελένα Μπονέρ, να γίνεται να τροποποιηθεί ο τίτλος του βραβείου και να μιλάμε για βραβείο Ζαχάροφ Μπονέρ. Θα ήθελα να πω ότι η Ελένα Μπονέρ δεν ήταν μόνο σύντροφος του Ζαχάροφ, προώθησε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πρώην Σοβιετική Ένωση και προώθησε την ανθρωπιστική, την, τα ανθρώπινα δικαιώματα, με συγχωρείτε, στην πρώην Σοβιετική Ένωση υποστηρίζοντας το έργο του συζύγου της. Και εξαιτία εργασία εργασίας της Ελένα Μπονέρ, η, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προβλήματα ως προς αυτά διαδόθηκαν διεθνώς και α, θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεται η κοινωνία των πολιτών και κατά πόσο μπορούμε να μετονομάσουμε αυτό το, γραφείο, το βραβείο, βραβείο Ζαχάροφ Μπονέρ. Ε, όχι μόνο για τυπικούς λόγους, αλλά και για ουσιαστικούς. Άλλα σχόλια ή παρεμβάσεις παρακαλώ. Συνάδελφε Ταβάρες, θα σας φέρουμε σε επαφή και με το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα έρθουμε σε επαφή με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να προωθήσουμε τη, τα θέματα αυτά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθεροτυπία, την ελευθερία του εκφράζεστε. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Monsieur le Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αλβάρ Μισατερή, είμαι αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ιράν, στην Ευρώπη. Το Ευρωκοινοβούλιο και ο ΙΕ πανηλημμένα έχουν καταδικάσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Είναι κρίμα λοιπόν που σήμερα δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνο εδώ για τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν που να είναι προσκεκλημένος. Ξέρετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ στο Ιράν, δύσκολη στο Ιράν, καταστροφική θα έλεγα. Κάθε μέρα κρεμάνε ανθρώπους, καταδικάζουν σε θάνατο, δέρνουν, μαστιγώνουν. Ε, προημερών η κυβέρνηση του Ιράν θέλει να αποφάσισε να δημιουργήσει ένα φίλτρο στο διαδίκτυο ε, ώστε η ενημέρωση στο Ιράν να περνάει από φιλτράρισμα. Υπάρχουν δύο αδελφοί ιατροί που αγωνίζονται στο Ιράν απλώς και μόνο για να ενημερώσουν τον λαό για το AIDS. Και λόγω αυτής της δραστηριότητας ε, φυλακίστηκαν για πέντε χρόνια καταδικάστηκαν σε φυλάκιση. Λοιπόν, αξίζουν το βραβείο Ζαχάροφ και πρέπει να τους προστατεύσετε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρέμβασή σας. Σας παρακαλώ. Να μην ε, ντρέπεστε, ζητήστε το λόγο. Δώστε μας τα παραδείγματα ενδεχομένως από τις χώρες σας. Εδώ είμαστε εμείς για να σας ακούσουμε. Δεν λησμονούμε όμως ότι ξαναρχίζουμε ακριβώς τις δύο. <clears throat> Έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Θέλετε εσείς να πείτε κάτι από το πάνελ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στην έκκληση που έγινε για τροποποίηση του ονόματος του βραβείου, του Ζαχάροφ δηλαδή. Έγινε αναφορά στην κυρία Έλενα Μπονέρ και υπόθηκε ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ε, δραστηριότητα του Ζαχάροφ. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτα, σαφε, ε, απόλυτα σωστό, γιατί ναι, συναντήθηκαν πολλές φορές μετά την ε, πρώτη απονομή. Ήταν ε, η κυρία Μπονέρ βεβαίω μέλος της Επιτροπής Υπερασπιστών των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, ήταν πολύ καλή φίλη της οικογένειας Ζαχάροφ και αξίζει ασφαλώς ε, να τιμάμε τη μνήμη της ίσως με ένα άλλο βραβείο διαφορετικό το να αλλάξει όμως όνομα το βραβείο Ζαχάροφ νομίζω δεν θα ήταν παραγωγικό φανταστείτε να αλλάξει όνομα το βραβείο Νόμπελ και ονομάζεται Νόμπελ Σφάιτσερ. Αποτελεί παράδοση πλέον το βραβείο Ζαχάροφ, έτσι ονομάζεται. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να μπορούμε να βρούμε υποστηρικτές, χορηγούς και ε, εφορευτική επιτροπή που θα στήριζαν ένα βραβείο Ελένα Μπονέρ, που θα ήταν βεβαίως εξίσου σημαντικό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ για την απάντηση και τις παρατηρήσεις σας. Αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου να πω μερικά λόγια, κλείνοντας αυτή την πρώτη μας ε, συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει βεβαίως το έργο του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε όλες μας τις εκθέσεις και σε όλα τα ψηφίσματα για κατεπήγοντα θέματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία επίσης πιστεύω καταγράφουμε αυτό το μέλημα. Και υπάρχουν βεβαίως δύσκολες υποθέσεις, πρέπει να υποστηρίζουμε πάντοτε αλλά δεν πρέπει και να λησμονούμε την κοινωνία των πολιτών στις χώρες σας. Πόθηκε δηλαδή, πολύ σωστά, ότι πρέπει οι λαοί οι ίδιοι στις χώρες αυτές να αλλάξουν την κατάσταση, να προξερήσουν την αλλαγή του συστήματος προς την ε, δημοκρατία, προς το στόχο της δημοκρατίας. Άρα χρειάζεται συνεργασία και συνεργασία μεταξύ όλων των ανθρώπων, των λαών, των εκατοντάδων χιλιάδων των πολιτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε εσάς στις χώρες αυτές, γιατί έτσι διευκολύνεται το δικό μας έργο σε κάθε προσπάθεια συνεργασίας που ξεκινούμε εσείς μας βοηθάτε. Συνεχίζουμε λοιπόν και τώρα το Δεκέμβριο είπατε εκπρόσωπος ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης η κυρία Άστον θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια αναθεώ, την έκθεση, έκθεση, την επισκόπηση καλύτερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ανά τον κόσμο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια έκθεση πολύ σημαντική για μα που θα συζητήσουμε με τον κειμενικό τρόπο εν ώψη και, της, και υπό το πρίσμα καλύτερα τη λειτουργία τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με του διπλωμάτε μα αφοσιωμένα εργάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και τα θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το δίκτυό μας, η δικτύωσή μας, δικτύωση δηλαδή του βραβείου Ζαχάροφ που επιτρέπει τη συνάντηση των τιμηθέντων με το βραβείο Ζαχάροφ είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας καθήκον. Και είμαστε βεβαίως ε, πρόθυμοι και περιμένουμε να γίνουν αντίστοιχε συναντήσεις και στο μέλλον. Θα μπορούσα να πω ίσως του χρόνου ή σε δύο χρόνια Πάντως το αργότερο σε δύο χρόνια θα πρέπει να ξανασυναντηθούμε. Είμαστε ευγνώμονες που βρισκόμαστε μαζί, που είμαστε μαζί. Διότι όπως υπόθηκε, εάν είμαστε μαζί, οπουδήποτε και αν είμαστε σαν άνθρωποι, αισθανόμαστε καλύτερα, αισθανόμαστε πιο ισχυροί, πολύ πιο ισχυροί από την ε, άποψη των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Θα σας ξαναδώ λοιπόν στις 2. Το βράδυ θα είμαστε στο Centrum Bozar με τη μεγάλη μας ε, συνεδρίαση, μεγάλη εκδήλωση, που θέμα έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή δικαιώματα της γυναίκας, γιατί ξέρουμε ότι ταυτίζονται οι έννοιες. Αλλά τα καλά νέα τώρα είναι ότι μπορούμε να πάμε για φαΐ. Χαίρετε.